Ελπίζω είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο την ε, συνεδρίασή μας. Ε, Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Έχουμε κάποια πραγματάκια πρωί-πρωί. Από τώρα μέχρι τις 11, δύο ώρες. Και μετά άλλες δύο ώρες το απόγευμα. 4 ε, και 45 με 6 και 45. Οπότε, Ξεκινάμε με τα γνωστά έγκριση ημερήσιας διάταξης, αλλά πριν από αυτό να ξεκαθαρίσω τα τεχνικά. Είναι η ένατη συνεδρίαση που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη. Έχετε λάβει τις τεχνικές πληροφορίες από τη γραμματεία. Σε περίπτωση προβλημάτων ενημερώστε μας για να υπάρξει κάποια τεχνική βοήθεια. Όσον αφορά τη διερμηνία υπάρχουν έξι γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, γερμανικά και ελληνικά. Και τα Ολλανδικά. Και παρακαλώ να μιλάτε τη γλώσσα σας αφού έχουμε διερμηνία και κατά τρόπον ώστε οι οι ε, να μπορούν να δουλέψουν. Και βεβαίως ζητάμε την κατανόησή σας και πάλι για τις τεχνικές δυσκολίες που έχουμε να ξεπεράσουμε ε, όταν μιλάμε για βιντεοδιασκέψεις. Λοιπόν, έγκριση ημερήσιας διάταξης, έχετε τα πρακτικά. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Μετά έχουμε κάποιες ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Συνήθως ανακοινώνουμε τον ορισμό εισηγητών. Έχουμε γνωμοδοτήσει Λένα Η εισηγήτρια για την έκθεση ΑΦΕΤ ΝΤΡΟΑ, έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλίας για κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά. 8 Ιουνίου 4 η ώρα το απόγευμα προθεσμία για τροπολογίες, ε, για ορισμό εισηγητών, λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση εγκρίνεται και μετά κάποιες πράξεις κατά εξοδότηση και κατά εφαρμογή. Υπάρχει ένα σχέδιο απόφασης της Κομισιόν 20 ε, Μαΐου για οικονομικές δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ταμείου Ασύλου και Ένταξης. Δεν είχαμε κάποια αντίρρηση. 12 Μαΐου επίσης λάβαμε το σχέδιο τροποποιητικής απόφασης ε, επί του κανονισμού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ζητήματα τελωνίων, ε, το οποίο το λάβατε όλοι μέσω του ενημερωτικού δελτίου, δεν λάβαμε κάποια αντίρρηση. Τώρα λοιπόν να σας πω ότι έχουμε και μια ψηφοφορία σήμερα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε όμως με το σημείο 4, κατάσταση στην ζώνη Σέγγεν μετά το ξέσπασμα του ιού COVID-19. Ε, την χάνει να είμαι ο εισηγητής, ως πρόεδρος. Οι βουλευτές που θα ψηφίσουν παρακαλούνται να το κάνουν με τον γνωστό τρόπο, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα όλες τις φορές. Έχετε το γνωστό email, τη γνωστή φυρίδα όπου μπορείτε να ψηφίσετε. Πρώτα απ' όλα θα δούμε αν υπάρχει απαρτία. Παρακαλώ λοιπόν την γραμματεία να με ενημερώσει αν υπάρχει απαρτία για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Καλωσορίζω και τους ε, παρόντες ε, στην αίθουσα. Παρακαλώ τους βουλευτές να πατήσουν το κουμπί της ομιλίας ε, όσοι είναι στο... στην τηλεδιάσκεψη για να ξέρουμε ότι έχουμε απαρτία και να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ε, υπάρχει απαρτία. Ωραία, σας ευχαριστώ που σηκώσατε το χέρι ή πατήσατε το κουμπί, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορείτε λοιπόν να τυπώσετε το ψηφοδέλτιο, συμπληρώνετε το όνομά σας, ψηφίζετε, συν, πλην ή μηδέν για αποχή, το σκανάρετε, το φωτογραφίζετε, στέλνετε την εικόνα, το υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο στη γνωστή θηρίδα και μόνο όσα έχουν σταλεί στο επίσημο email του Κοινοβουλίου θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας η οποία ξεκινάει τώρα θα ανακοινωθούν στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Το απόγευμα λοιπόν. Έτσι θα ξέρουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Περνάμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Ίνετφελντ, κύριε Πρόεδρε, θέλει να πει κάτι από τις διαδικασίες. Ήθελα να θέσω κάτι στην αρχή στις ε, αρχικές σας παρατηρήσεις, αλλά είναι δύσκολο όταν κάποιος είναι εντός της αίθουσης ε, να προσελκύσει την προσοχή σας. Όταν αναφέρατε τις γλώσσες, να τονίσω ότι υπάρχει ένα θέμα με τους διερμηνείς, τους ελεύθερους επαγγελματίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διοίκησή μας, εξ ονόματος μας, ακύρωσε τα συμβολεά τους βασικά έχουν μείνει χωρίς καμία προστασία, δεν έχουν καμία οικονομική στήριξη γιατί δεν καλύπτονται ούτε από το βελγικό σύστημα ούτε από το σύστημα της Ένωσης. Είναι έσχος να μεταχειριζόμαστε έτσι ε, ανθρώπους τους οποίους χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχουν, έχω επικοινωνήσει μέσω διαφόρων διάβλων, αλλά φαίνεται ότι ο Γενικό Γραμματέα έχει άλλε δουλειέ. Ελπίζω λοιπόν να το θέσετε και στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ε, με του Προέδρου των Ομάδων, γιατί νομίζω το οφείλουμε στου ανθρώπου οι οποίοι θα επανέλθουν μετά την κρίση και αναμένουμε από αυτού να συνεχίσουν να εργάζονται ε, και ε, συνήθω και πέρα από το ωράριό του. Σας ευχαριστώ κυρία Ινετφέλντ για το θέμα το οποίο θέσατε. Είναι πράγματι ευαίσθητο. Σίγουρα κάποιοι από εμά δεν γνωρίζαμε την κατάσταση την οποία αναφέρατε. Οπότε είναι χρήσιμο το να το θέσετε γραπτός για να μεταφέρουμε το μήνυμα. Οπωσδήποτε και άλλες επιτροπές έχουν τις ίδιες ανησυχίες με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζητάω εσείς να το κάνετε γραπτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε είναι προσωπικό μου ζήτημα. Είναι ε, δουλειά του Κοινοβουλίου. Ναι, ναι, το γνωρίζω, το ξέρω πως δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Αφορά πράγματι τις ε, συνθήκες εργασίας ε, κάποιων ανθρώπων. που εξαρτώνται από αποφάσεις που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταφέρουμε οπωσδήποτε τις ενισχύσεις. Απλά να πω βεβαίω ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους διερμηνείς στη δική μας επιτροπή, αλλά σε όλες τις επιτροπές. Οπότε θα θέσουμε το θέμα στην ε, διάσκεψη των πρόεδρων και των πρόεδρων των επιτροπών για να δούμε την ε, κατάσταση. Αυτό, αυτό έλεγα. Και το σημειώνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο ουσιαστικό θέμα. Έχουμε πτυχές ε, δεοντολογικών ε, θεμάτων ε, της τεχνητής νομοσύνης, ρομποτικής λοιπά Έχουμε την κυρία Κάνκο, την εισηγήτρια από το ECR και αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Κάνκο θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης για να το εξετάσουμε. Θα λάβει τον λόγο πρώτη. Προτείνω 7 λεπτά και μετά μπορούμε να περάσουμε στους σκιώδεις εισηγητές. Ένας από κάθε ομάδα. 20 λεπτά έχουμε προγραμματίσει για αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι αρκούν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Κάνκο. Έχετε τον λόγο. Good morning and thank you very much, Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο μας σε αυτό το μέτωπο για ρομποτική, σχετικές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που προσφέρονται από αυτές τις τεχνολογίες για οικονομία και κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, όπως κάθε με τεχνολογία, θα πρέπει να δούμε ότι όπου υπάρχει καινοτομία θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Και Κάτι που πάντοτε ξεκαθαρίζουμε είναι ότι θα πρέπει τα δικαιώματα να συμβαδίζουν με την ασφάλεια. Αυτά όσον αφορά την δικαιοσύνη, μια που είναι θέμα και δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων, οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τα φροντίσουμε και να είναι ασφαλέστεροι οι πολίτες. Οι μεγάλες εταιρείες του ίντερνετ, ε, αυτοί που έχουν το τεχνολογικό νέφος θα πρέπει αυτά να τα φροντίσουν. Μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει για τη φύλαξη των συνόρων, μπορεί να βοηθήσει καταπολέμηση τρομοκρατίας και αντιμετώπιση επιγουσών καταστάσεων. Προσέξουμε την προσερτητικού βίου και τις πολιτικές ελευθερίες. Στα λάθος χέρια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παροξύνει τις ανισότητες κοινωνικές, μεταξύ φίλων, τον ρατσισμό. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές, ένα στεγανό πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Μάθαμε από τον κανονισμό για την πρόσταση των δεδομένων ότι πρόκειται για δύσκολο έργο και θα πρέπει να υπάρξει θέσπιση κανόνων εκ των προτέρων. Ακόμα και όταν είναι κανόνες ενδοτικού δικαίου και αυτό να γίνει επαναλαμβάνω νωρίς. Αυτό να αφορά το design της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Να υπάρχει αναλογικότητα να υπάρχει κάποιο είδους διαφάνεια και τρόποι για να υπάρχει έλεγχος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται ισχύουσα νομοθεσία και για την συλλογή αλλά και αποθήκευση δεδομένων για όλους τους ε, τομείς, πανεπιστήμια, ε, νομικούς, ε, επιστήμονες, μηχανικούς, ένα πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έχουμε δει τόσα έργα που με τους ε, υπολογιστές καταπολεμείται το έγκλημα. Αυτό ήταν επιστημονική φαντασία και τώρα είμαστε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Άρα να σιγουρέψουμε ότι μπορούμε νομοθετικά να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Με αυτή μου τη γνωμοδότηση αυτό θέλω να υλοποιήσουμε βασικές αρχές από πλευράς αρμοδιοτήτων μας, ασφάλεια, δικαιώματα και ελευθερίες. Ακόμη υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλω να προσθέσω που δεν μπόρεσε λόγω των τρεχόντων περιορισμών. Είναι τα ζητήματα αυτά περίπλοκα, πρέπει να μας προβληματίσουν, να τα διερευνήσουμε. Οπότε θα υποβάλω και άλλες τροπολογίες για το κείμενο που έχετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η παραπληροφόρηση, η ηγετική πρωτοπρόθεση της Ευρώπης, όλα αυτά να είναι ζητήματα που αναλαμβάνουν υπόψη τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ τους ε, σκιώδες εισηγητές και περιμένω τη συνεργασία τους για να γίνει το κείμενό μας όσο γίνεται πιο ενδιαφέρον. Πάντοτε ε, είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας. 11 Ιουνίου Τέσσερις ώρε είναι η προθεσμία τροπολογία. Στις 23 Ιουνίου θα τα συζητήσουμε με τους ε, ηγητές, να έχουμε όσο γίνεται πιο δυναμικό κείμενο και να μπορούμε να έχουμε προσθέμενη αξία στο έργο της Επιτροπής μας. Και ευχαριστώ φυσικά και την ε, γραμματεία. Περιμένω τα σχόλιά σας, τη συνεργασία μαζί σα. Thank you, for your presentation of your draft opinion. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας όσον αφορά ρομποτική, σχετικές τεχνολογίες, όσον αφορά τις διοντολογικές πτυχές. Και τώρα έχουμε τους σκιώδες. Πρώτα-πρώτα για το Αλγικύρους Πέτερ. να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε και φυσικά προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Είναι απλή η επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Να αναπτύξουμε λοιπόν την ε, τεχνητή νοημοσύνη ή... και να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές ή να ακολουθήσουμε τελικά την, ε, τη ΣΥΠΑ και την Κίνα χωρίς τα οικονομικά ωφέλη. Θα πρέπει να είναι σαφές λοιπόν ότι οι πρωτοβουλίες μας λοιπόν θα πρέπει να έχουν συνέχεια, διασφαλίζοντας τις αξίες μας. Και θα πρέπει όλα αυτά φυσικά να αντιμετωπιστούν με ένα λογικό τρόπο. Για το σκοπό λοιπόν αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό αλλά και ευέλικτο πλαίσιο. Προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προωθηθούν. Και θα πρέπει να υπάρξει και μια σωστή αξιολόγηση κινδύνου. Έχω κάποιες προτρήσει να κάνω. Και φυσικά θα τα συζητήσουμε αυτά και με την εισηγητρία, αλλά να αναφέρω κάποια στοιχεία. Δεν μου αρέσει αυτό το ethical by default, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια, ένα σωρό ε, ομπρέλα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δεντολογικό ε, εξορισμού. Ethical by default. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν το σχετικό πλαίσιο. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέμα των επιρροών και τη ευθύνη. Ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικό για την Επιτροπή μα, Ωστόσο, θα πρέπει να κοιτάξουμε και πέρα από την δικαιοσύνη τον τομέα της δικαιοσύνης. Αν δεν τα ορίσουμε όλα αυτά, θα υποστούν πιέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από το πλαίσιο της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το θέμα της αναλογίας. Για να διατηρηθεί η οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων και να υπάρχει πλήρης ευθύνη από τα κρατη θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα αυτά με έναν κανονισμό για την ευθύνη που φέρουν οι παραγωγοί ε, τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί κάπου στο κείμενο. Κατά τέταρτον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη να μην υπάρχει μεροληψία σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση προσώπου. Ακούσαμε τι σημασία έχει αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εφαρμογή ε, της δικαιοσύνη ε, και μας μίλησε και η αστυνομία του Σικάγο για τα θέματα αυτά τον Φεβρουάριο. Γιατί ο ρατσισμός μπορεί να κατοχυρωθεί ουσιαστικά με τέτοιου τρόπου στην κοινωνία και να υπάρξει αυτόματη διακριτική μεταχείριση. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Πάση θυσία. Τέλος, το οντολογικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει για όλους. Όλους όσοι σκοπεύουν να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και θα πρέπει να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτερς, ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε στον σκιώτη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, την κυρία Κατερίνα Βαρλάιν Καλημέρα σας και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κάνκο για το σχέδιο γνωματότησης αυτό, για το πολύ συναρπαστικό αυτό θέμα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία και θα αλλάξει σε κάθε περίπτωση το τοπίο της ζωής μας, σε κάθε έκφανσή του. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί, αλλά χρειάζεται και να ρυθμιστεί. Και υποστηρίζω πολλά από αυτά που η κυρία Κάνκο σε ό,τι αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία και να προστατεύει τους πολίτες. Και να πρέπει, θα πρέπει να σέβεται και την αρχή του να εξηγείται σωστά. Θεωρώ ότι κάποιε πτυχέ θα μπορούσαμε να τι εξετάσουμε λίγο πιο ανταλλαχώ. Θα θέλαμε λίγο πιο ακριβή διατύπωση, έναν πιο φιλόδοξο κανονισμό σε κάποιε περιπτώσει και θα επικεντρωθώ σε τέσσερα θέματα. Καταρχάς, θα πρέπει να ορίσουμε τι θα πρέπει να περιέχει αυτό το δεοντολογικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να αποτρέπεται οποιαδήποτε μορφή διακριτική μεταχείριση ε, από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για σεξουαλικό προσανατολισμό, εθνότητα, ε, θρησκεία, φύλλο, ε, οτιδήποτε. Δεν θα πρέπει να παίζουν ρόλο στους αλγοριθμούς και οποιαδήποτε μεροληψία θα πρέπει να αποτραπεί. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει και μια σκληρή ρήτρα για την αξιολόγηση, γιατί αξιολόγηση κινδύνου όσο πιο μεγάλος αντίκτυπος είναι ο αντίκτυπος του κανονισμού, τόσο πιο μεγάλη, το μεγάλο έλεγχο χρειάζεται. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά έναν αργόριθμο ο οποίο αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν σωστό έλεγχο. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τον τομέα τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση της Ιβάνα για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν α, κοινά κριτήρια για να υπάρχει δεντολογική συμμόρφωση. Και τμήμα της πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανωνυμοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης αλγοριθμών. Και θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει και αυτή η εταιρική ψηφιακή ευθύνη, όπως αποκαλείται. Να υποστηρίξουμε δηλαδή τις επιχειρήσει εκείνης που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με δεντελογικό τρόπο. Και έτσι μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα διάχυθουν στην αγορά εργασίας. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια σωστή γνωμοδότηση για την εντολογική αυτή διαμόρφωση των ε, τεχνολογιών και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας τις επερχόμενες συναντήσεις των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να ακούσουμε τους σκιώδεις ε, των Ρενιού. Ο κ. Τουντουράτσε, σας ευχαριστώ. Το οντολογικό πλαίσιο για την ε, τεχνητή νοημοσύνη είναι προφανώς ένα θεμελιώδες στοιχείο στη στρατηγική μας και στο όραμά μας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ως Ρενιού το έχουμε πει αυτό ξεκάθαρα στο έγγραφο τοποθέτησή μας φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω διευκρίνησε τη σχετική στρατηγική το Φεβρουάριο και άρα θεωρώ ότι είναι λογικό το ότι εξετάζουμε αυτή την πτυχή. Συμφωνώ με την γενικότερη κατεύθυνση την οποία έχει ακολουθήσει η συγγητρία. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις, ωστόσο, τις οποίες έχουν επισημάνει και στην αδελφή. Όπως, για παράδειγμα, η ανάγκη διαφοροποίησης. Είτε πρόκειται για αξιολόγηση κινδύνου, είτε πρόκειται για διαφοροποίηση. Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια νομοθεσία τα καλύπτει όλα σε ό,τι αφορά τα δοντολογικά πρότυπα, γιατί υπάρχουν ε, τέτοιες τεχνολογίες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, αφορούν τη ζωή του ανθρώπου και χρειάζεται λοιπόν εδώ πιο προσεκτική ρύθμιση, να μην υπάρχει ημεροληψία, αντικριτική μεταχείριση στον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογιών αυτών. Από την άλλη, υπάρχουν και αλγοριθμοί οι οποίες οι οποίοι καθορίζουν, ε, για παράδειγμα, πώ λειτουργεί μια μηχανή μέσα σε μια υποθήκη. Εκεί πέρα τα χρειάζονται ιδιαίτερα δεντρολογικά πρότυπα και άλλε τέτοιε τεχνολογίε στη βιομηχανία, οι οποίε θα πρέπει να έχουν περιθώριο να αναπτυχθούν και να προωθηθούν για να ενισχύσουν την οικονομική μας θέση. Εδώ χρειάζεται λοιπόν ε, διαφοροποίηση, αξιολόγηση κινδύνου και οι τροπολογίες τις οποίες θα προτείνω μέχρι την επόμενη εβδομάδα ακριβώς αυτό το στόχο θα έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Tudorachi. Let's move to ID. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στον ε, σκιοδησηγητή της ομάδας ID. Δεν είναι συνδεδεμένος από ό,τι φαίνεται. Οπότε πάμε τώρα στον κύριο Λαγκουντίνσκι από τους Πράσινους. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και σας και τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το ενδιαφέρον αυτό σχέδιο έκθεση. Ελπίζω να μπορέσουμε να το διευρύνουμε. Υπάρχουν τέσσερα σημεία που είναι σημαντικά για εμάς. Κάποια ήδη αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα η λεπτή ισορροπία μεταξύ καινοτομία αφενός και ανθρωπίνων δικαιωμάτων απ' την άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Σαφήνεια επίσης των ενιών επί των οποίων ε, εργαζόμαστε είναι κάτι το σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες ε, τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι όλες όριμες ε, ούτε είναι ήδη υπάρχουσες για να εκτεθούμε στους κινδύνους που κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι μας εκθέτουν. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ακριβώ το τι εννοούμε και κάτι άλλο ο, ο ρόλος ε, της νομικής ρύθμισης. Η ιδεολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα δικαιώματα βάσει του νόμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να υποκαθιστούμε ε, σαφή ε, δικαιώματα από δεοντολογικούς κώδικες. Οι δεοντολογικοί κώδικες, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πρόσβαση, να μπορεί κανείς να προσφύγει ε, επίσης ε, κατά ε, διακριτικής μεταχείρισης και θα πρέπει να δούμε και το πώς θα μπορέσουν ακριβώς να μεταφραστούν θεσμικά αυτά. Υπάρχει ήδη μια πρόταση για μια υπηρεσία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δημιουργήσουμε άλλη μια υπηρεσία ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια που έχουμε, αλλά κάποιος ε, θα μπορούσε να επιβλέπει ε, αυτά τα πράγματα. Οπότε ας ε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Λαγκουντίνσκι. Τώρα, ο, Κυρία Κλέρ Ντέιλι από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Όπως είπε, είναι περιορισμένη ε, λόγω των συνθήκων και έχουμε κάποιες διαφωνίες αλλά όχι ουσιαστικές. Ε, λοιπόν, σε ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα στα οποία έχουμε διαφωνίες είναι το θέμα το οποίο αφορά την χρήση τεχνητής νοημοσύνης ε, στο σύστημα ποινική δικαιοσύνη. Και δεν θα μπω τώρα στις ε, λεπτομέρειες. Για εμάς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει η υποδομή ε, που θα αφορά ε, πολλούς τομείς, από την εκπαίδευση, την υγεία, τις μεταφορές ε, κτλ. Οπότε το ποιος θα έχει και θα ελέγχει αυτήν την τεχνολογία, το ποιος θα τη χρησιμοποιεί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπως είπε και ο Πούτιν, οι... αυτοί οι οποίοι έχουν την ιδιοκτησία και τον έλεγχο θα έχουν τον κόσμο και βεβαίως Έχουμε εδώ πέρα αμερικανικές και κινέζικες εταιρείε, οι οποίες ξοδεύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα, δηλαδή το πώς θα έπρεπε να είναι υποδημόσιο έλεγχο αυτή η τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανισχύει και εδώ πέρα συμφωνώ με τον συνάδελφο από τους πράσινους. αυτού είμαστε εδώ πέρα και μιλάμε για ένα βήμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμισής, αλλά δεν μιλάμε για νομοθεσία, αλλά για ε, κανόνες δεοντολογίας και μας λέτε η νομοθεσία θα έρθει αργότερα. Αυτά όμως είναι κάπως αφηρημένα ως προς το τι θα γίνει. Το μόνο το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής είναι κώδικες δεοντολογίας. Δεν επαρκεί. Δηλαδή και Αμερικανική αστυνομία έχει υπογράψει για πράγματα, αλλά αυτό δεν του εμποδίζει να ρίχνει δακρυγόνα σε διαδηλωτέ ε, κτλ. Και μιλάμε εδώ πέρα για εταιρείε οι οποίες είναι μεγαλύτερε από κράτη και φτάνουν σε κάθε πτυχή της ε, ζωής ε, των πολιτών. Και έχουμε εδώ πέρα, τα... δηλαδή θα αρκεστούμε στο ότι η Google λέει δεν είμαστε κακοί. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι Καλά είναι όλα αυτά, αλλά να μην ε, χάνουμε ακριβώς ε, τα γεγονότα. Η Google έχει ξοδέψει 8 εκατομμύρια για lobbying εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οπωσδήποτε θα είναι πολύ ικανοποιημένοι με έναν κώδικα διοντολογίας. Οπότε καλό είναι να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλοι ευχαριστούμε τους κοιόδης συζητητές. Πριν επιστρέφουμε στην κυρία Κάνκο, νομίζω ότι ο κύριος Σαθαλέρος θέλει να παρέμβει για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα, όπου έχουμε μια σημαντική συζήτηση. Κύριε Θαρθαλέχος, είστε εκεί? Sir, um, you have deactivated your camera and you are online. You can... Είστε συνδεδεμένος. Μπορείτε να μιλήσετε. Could you please connect your camera? Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερά σας. at the beginning of this session, of course, just... Στην αρχή της ε, συνεδρίασης ε, είχα ζητήσει την κατανόησή σας, λέει ο Πρόεδρος, για τις ε, δυσκολίες που έχουμε συνήθως με αυτές τις συνδέσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Ε, συμβαίνουν αυτά. Προφανώς ο κύριος Θαρθαλέχος προσπαθεί να συνδεθεί, αλλά δεν είναι δυνατόν. Ε, λοιπόν, κύριε Θαρθαλέχος, πρέπει να προχωρήσουμε να επανέλθουμε στην εισηγήτρια, στην κυρία Κάνκο, να κάνει τις ε, τελευταίες της παρατηρήσεις και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα σας τα σχόλια. Συμφωνώ πλήρως ε, με το ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ε, λεπτομέρειες, αλλά όπως είπαμε ήδη, αυτό ήταν περιορισμός ε, λόγω του αριθμού λέξεων που έχουμε ε, κάτι το οποίο βέβαια μας απογοήτευσε γιατί είχαμε μεγαλύτερο κείμενο και ε, μας δυσκολεύει αυτή η υπόθεση γιατί η δουλειά μας βεβαίως συνεχίζει και πρέπει να μπορούμε να την κάνουμε αποδοτικά. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει Μπορούμε να δεχτούμε τροπολογίες και συμβαστικά κείμενα. Επίσης πρέπει να εστιάσουμε στις αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής μας. Πολιτικές ελευθερίες, θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου. Δηλαδή, δηλαδή αν ε, ξεφύγουμε από αυτά δεν ε, θα μας βοηθήσει πολύ. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ να αποτελούν πηγή έμπνευσης. We Σας ευχαριστούμε κυρία Κάνκο. Και ε, με συγχωρείτε για το ότι δεν μπόρεσε να συνδεθεί ο κύριος Θαρθαλέχος. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει μέχρι τις 11 μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Το σημείο παριθμών 5. Αντίκτυπος του COVID-19 της πανδημίας στην κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Θα ακούσουμε τον κύριο Γκουζντελ του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την τοξικομανία και τα ναρκωτικά στην Λισαβόνα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας ad hoc ε, που έχει κάνει η υπηρεσία αυτή για να αναλύσει τον αντίκτυπο του COVID ε, της πανδημίας ε, στο θέμα των ναρκωτικών. Θα κάνει μια παρουσίαση και μετά θα δεχτεί ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές από κάθε πολιτική ομάδα που ε, θα θέσουν ερωτήσεις στον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ας ακούσουμε όμως την ε, παρουσίασή του. Κύριε Γκουσδέλ, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουμε κάνει για τον αντίκτυπο του COVID-19 στο θέμα των ναρκωτικών. Πρώτα απ' όλα... Και να διευκρινίσουμε ότι τίθεται και το θέμα της επίδρασης του COVID από πλευράς ε, των, ε, της χρήσης ναρκωτικών ε, των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά και στην ε, αγορά ναρκωτικών. Δεν πρόκειται για αξιολόγηση της επιδημίας σε όλα τα στοιχεία της κατάστασης, γιατί καταρχά είναι πάρα πολύ νωρίς και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία και με άλλες ε, ε, οργανώσεις, την Europol, την CDC, για να δούμε τι γίνεται. Προσαρμόσαμε λοιπόν το σύστημα συλλογή δεδομένων σε ό,τι αφορά τα νέα προβλήματα για μια πιο ασφαλή Ευρώπη και κάναμε νέες ασκήσεις συλλογής δεδομένων με γρήγορο τρόπο και νέες μελέτες. Μία μελέτη στο διαδίκτυο, χωρίς να ξεχάσουμε, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά και το Darknet. Και σε ό,τι αφορά την κοινή έκθεση MCDC και MA, Europol για την επίδραση του COVID. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στα στοιχεία αυτά και κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήταν ε, και πριν εξαιρετικής σημασίας και παρέμειναν μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά το σύστημα έγκρισης προειδοποίησης, σε ό,τι αφορά τις ε, ουσίες, τις επικίνδυνες ουσίες. Όπως ξέρετε, έχουμε τις νέες αυτές ουσίες, οι οποίες ονομάζονται ίσω των Ινανίνες, μια νέα ομάδα ουσιών έγινε αξιολογήση κινδύνου την προηγούμενη εβδομάδα, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθούμε τις ε, αποφάσεις. Ποιες ήταν λοιπόν οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τη χρήση ναρκωτικών. Καταρχάς, διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές που προκλήθηκαν από την επιδημία είναι διαφορετικές ανάλογα με την ουσία, ανάλογα με την κατηγορία, αλλά και τη χρήση της ουσίας. Καταρχάς, λοιπόν, το συγκείμενο είναι πιο σημαντικό παραποτέ. Και σε κάποια η χρήση της κάναβης ενδεχομένως να παρατηρήσαμε συγκέντρωση ουσιών από τους χρήστες εν ώψη του lockdown. Αλλά και λόγω των μέτρων του lockdown ήταν πιο εύκολο, ήταν πιο δύσκολο να κυκλοφορήσει η κάναβη από τη μία χώρα στην άλλη και έτσι μειώθηκαν τα αποθέματα στους χρήστες. Δεύτερον, αύξηση της χρήσης αλκοόλ και φαρμάκων όμως. Εδώ να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στις βενζονδιαπίνες. Τέλος, φαίνεται ότι υπάρχει μία μικρή μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατά τη διάρκεια του lockdown σε αυτά τα φάρμακα που αποκαλούνται φάρμακα πάρτι. Κοκαίνη, έκσταση, ε, MDMA, αμφεταμίνες. Αυτή η αλλαγή όμως δεν ήταν και δραματική. Και δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί και αυτή η τάση, η μειωτική, μιας και η ζωή σιγά σιγά επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα και οι δραστηριότητε οι ανθρώπινε επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχουν λοιπόν νέα είδη χρήση και νέοι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν. Μεγαλύτερη κίνδυνη και μεγαλύτερη έκθεση για κάποιες ομάδες. Να σας περιγράψω λοιπόν τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τον κύκλο χρήσης ε, ναρκωτικών και να περάσω στην κατάσταση τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά. Να ξεκινήσω αναγνωρίζοντας τη σημασία των ε, ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της υγείας, που έδωσαν τόσο μεγάλη κατέβαλαν τόσο μεγάλες προσπάθειες χωρίς να έχουν σωστή, σωστές συνθήκες εργασίας απαραίτητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε και να ενταχθούμε για να είμαστε καλύτεροι και καλύτερα προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημία ή σε ενδεχόμενη μελλοντική πανδημία. Ένα λοιπόν βασικό μάθημα το οποίο πρέπει να εξαγάγουμε ω συμπέρασμα είναι ότι όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα τη υγεία θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε εξοπλισμό ασφαλείας και εξοπλισμό προστασίας από το COVID. Άρα βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο αντικτύπο στην κοινότητα των ε, ατόμων αυτών που φροντίζουν τους άλλους. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το χρόνο εργασίας. Το πρόβλημα λοιπόν που το ότι τα... Το πρόβλημα ήταν λοιπόν ότι τα κέντρα παροχής ε, υποστήριξης σε εξαρτημένους ανθρώπους δεν θεωρήθηκαν θεμελιώδεις υπηρεσίες. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε πραγματικά τα άτομα που δουλεύουν εκεί πέρα για το γεγονό ότι υπήρξε κάποια συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σε εξοπλισμό προστασίας από το COVID για την προστασία δηλαδή του προσωπικού σε περίπτωση ατόμων τα οποία είχαν προσβληθεί ενδεχομένω από το COVID. για να υπάρξει προστασία τους από έκθεση στον ιό. Και είχαμε και πολύ καλές εμπειρίες σε τοπικό επίπεδο πιο πολύ και όχι τόσο πολύ σε επίπεδο εθνικών στρατηγικών σε ό,τι αφορά την ανάγκη καινοτομίας, ευελιξίας εδώ έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα να επιδείξουμε. Και σε μια χώρα και πόλη όπως η Αθήνα, οι αρχές με την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων κατάφεραν να ανοίξουν ένα νέο καταφύγιο για όσους ήταν οι πιο ευάλωτοι σε ό,τι αφορά τη χρήση ναρκωτικών και ουσιών αύξηση λοιπόν ε, διαπιστώνουμε και της χρήσης των ε, τεχνολογιών εξ απόστασης ε, βιντεοδιάσκεψης σε κάποιες περιπτώσεις με τους ασθενείς. Κάτι εντελώς καινούριο ανήκουστο μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Αποτέλεσε μια ευκαιρία για μεγαλύτερη ευελεξία για κάποιες θεραπείες, ή τμήματα της θεραπείας οι οποίες μπορούσαν να καλύψουν κάποιες καινούργιες ε, ανάγκες που προέκυψαν αναπαντήχες. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε κάποιες πόλες, πόλεις διαπιστώθηκε μεγάλη μείωση των καταλόγων αναμονής. Επίσης ε, υπήρξε πρόκληση ε, για τις νέες αιτήσει όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνει σωστή αξιολόγηση και ο κανονικός προκαταρτικός έλεγχος όπως ηθίστε. Και νέε ανάγκε για τους πιο περιθωριοποιημένους πελάτες. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε ε, να δοθούν ε, υπηρεσίες, για παράδειγμα, για να πληθούν τα ρούχα των ανθρώπων αυτών και να τους πάμε τρόφιμα ε, νερό. Άρα, συνολικά διαπιστώνουμε ότι υπάρξει, υπήρξε μεγάλο, μεγάλη καινοτομία. Πολλές καινούργιες ε, διαστάσεις. Είναι καλή λοιπόν η στιγμή να διδαχτούμε από τα μαθήματα του COVID και να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι στα κρατημέλια αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες και όλα αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο στην αγορά των ναρκωτικών, διαπιστώνουμε ότι η λαθρεμπορία ναρκωτικών συνεχίστηκε μέσω των συνηθισμένων οδών παρά τον COVID-19 ή οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω του COVID κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε μειωμένα αποθέματα, αλλά βλέπουμε ότι η αγορά ήταν πάρα πολύ ανθεκτική τελικά και πολύ εφευρετική. Υπήρξαν, ε, υπήρξε αντικτύπωση λόγω του κοινωνικού τη κοινωνική αποστασιοποίηση, αλλά και εδώ οργανώθηκε μια χαρά η αγορά. Και γενικά λοιπόν και η μεταφορά άμα προσαρμοστήκε και τα μοντέλα αποστολής. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, είχαμε κατασχέσεις ναρκωτικών που είχαν, ε, για παράδειγμα, κρύφτη σε μάσκες οι οποίες μεταφέρθηκαν ε, στην Ευρώπη. σε ό,τι αφορά τα precursors. Και εδώ έχουμε περιορισμένες ενδείξεις για ελλείψεις αλλά δεν σταμάτησε η παραγωγή αμ, συμφετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη. Έχουμε κάποιες ενδείξεις. ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, αλλά δεν σταμάτησε η παραγωγή. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Ένας, ε, μία από τις προκλήσεις λοιπόν για τους επόμενους μήνες θα είναι να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις ε, και θα υπάρξει πραγματικά τεράστια αύξηση στην διαθεσιμότητα των ουσιών αυτών. Αν δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες. Καταρχάς, αυτό που μας απασχολεί είναι ότι το τοπίο επικοινωνιών έχει αλλάξει. Οι διαπροσωπικές ε, επαφές μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών έχουν αντικατασταθεί μέσω των ψηφιακών οδών και αυτό μπορεί να συνεχιστεί ω τάση και στο μέλλον. Και τέλος, ε, ε, επίσης, όλη η οικονομία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και οι δυνατότητες ε, ελέγχου και επιτήρησης. Επίσης, ε, οι προοπτικές διαφθοράς λόγω της ρίκνουσης της οικονομίας που αναμένεται. Και θα υπάρξει ενδεχομένω απόπειρα να παράγονται τα ουσίες αυτές πιο κοντά στον τόπο κατανάλωσης το μήνυμα που έχουμε λάβει και από τους επαγγελματίες του κλάδου και από τους πελάτες είναι ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως ήταν ε, εντελώς αναπάντεχες, τις οποίες ε, σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να συζητούσαν επί χρόνια και τώρα επιτέλους πέρασαν. σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λέγαμε ότι τίθεται ε, και θέμα φροντίδας και όχι επιβολής τιμωρίας. Αυτό ενδεχομένως να το καταφέραμε και λόγω της πανδημίας να το πετύχουμε. Παράλληλα το συζήτησαμε εδώ και καιρό. Μία δεύτερη πρόκληση από πλευράς δημόσιας υγείας. Την ανέφερα ήδη. Να εξετάσουμε όλα τα προγράμματα ε, ελέγχου χρήσης ουσιών ως τμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υπάρχει ίδια πρόσβαση σε αυτά. Και ενδεχομένω ε, στην πανδημία COVID, ε, μετά την επιδημία του COVID, να υπάρξει μεγαλύτερη ευαλωτότητα, καθότι θα είναι δύσκολο και από οικονομική άποψη η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Τρίτη πτυχή να υπάρξει μία σταθερή αντιμετώπιση των ναρκωτικών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Σε ό,τι αφορά και τους πόρους που διατίθενται για τις πιο ευάλωτες ομάδες που θα υποστούν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με άλλες ομάδες ανθρώπων οι οποίες λίγο πολύ είναι ακόμα ενσωματωμένες στην κοινωνία και θεωρώ θα δούμε κάποιες εξελίξεις στην αγορά εργασία, στην αγορά ναρκωτικών και θα πρέπει να τις παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου την Επιτροπή σας για την διαρκή υποστήριξη που μας δίνετε. Για μένα μία είναι η λέξη κλειδί. Και αυτό το είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές οικονομικο πλαίσιο. Και αυτή η λέξη είναι σημαντική, ιδιαίτερως μετά την πανδημία. Η ε, πρόταση για τον προϋπολογισμό του η MCDD, δυστυχώ θα πρέπει να διαπιστώσω ότι δεν συνάδει με την προτεραιότητα που δίνεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη μελλοντική πανδημία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 1,5 εκατομμύριο ή το 2021 και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η πρόταση αυτή όχι μόνο δεν είναι βιώσιμη, αλλά καθώς ο προπολογισμός για το 2021 ενδεχομένως να προσαρμοστεί μελεθνικά για το μελλοντικό πουδουπού, τελικά θα καταλήξουμε στα επόμενα χρόνια, αντί να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς όλους, ενδεχομένως να χρειαστεί να περικόψουμε αυτές τις υπηρεσίες που δίνουμε Θέλουμε λοιπόν μια δίκαιη αντιμετώπιση και βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ευχαριστεί τον κύριο Χόφτελ για το έργο του, αλλά και για την εισήγησή του. Μας παρουσιάσετε σύντομα όλα τα σημαντικά στοιχεία και τώρα να κάνουμε την ανταλλαγή ε, απόψεων. Πρώτα-πρώτα έχουμε τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Δύο λεπτά έκαστος. Και έχουμε και δεύτερο γύρο με συνέντευξη που θα θέλουν να μιλήσουν. Όπως πάντα πρέπει να τελειώσουμε μια που πρόκειται για τηλεσυνεδρίαση με ακρίβεια όποτε προβλέπετε. Οπότε, παρακαλώ να προσέξετε το χρονικό πλαίσιο Ξεκινούμε για αυτόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με την κυρία Λένα Ντυπών. Έχετε το λόγο. Η κυρία Ντυπών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόφς Ντέιλ για τα όσα μας εξήγησε. Ε, βέβαια, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα τώρα, οπότε πάλι καλά που τα κατάφερε. Να δούμε τι γίνεται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ε, αυτό σταμάτησε με την πανδημία, αλλά όχι για όλα. η Ηρωίνη, κοκαίνη, ακόμη, ακόμη ε, του συνήθες διάβλους φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, για πετε μας, το κέντρο παρακολούθησης έχει κάποια στοιχεία σε σχέση με κατανάλωση αυτών των σκληρών ναρκωτικών ε, ως προς ε, τα μέτρα, τα περιοριστικά μεγάλωσε σε κατανάλωση τρόφων όσον αφορά την ε, διανομή. Ε, ξέρουμε ότι λόγω της ε, πανδημίας η κατάσταση γίνει πιο δύσκολη. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιείται έχει η υπηρεσία σας ήδη συνεργαστεί με την Europol, με εθνικές αρχές, για κάποια εργαλεία λογισμικού. Δηλαδή, ακριβώς για το εμπόριο των ναρκωτικών, αλλά και για τους τελικούς χρήστες. Τι γίνεται. Μήπως κάποιοι τρόποι καινούργοι εμπορίου ναρκωτικών χρησιμοποιηθούν και μετά την πανδημία. Ακούσαμε τι είπατε για τους νέους, είπατε ότι έχουν περισσότερη βία, ε, ασταθής κατάσταση στην αγορά και ε, υπήρχε πρόβλημα για το πώς θα εντοπίσουν διοικητικές αρχές. Έχετε κάποιο οργανωμένο τρόπο, κάποια στρατηγική να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση για καταπολέμηση των σχετικών δικτύων. Thank you. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Ντυπών. Και τώρα, σοσιαλιστές. Η Κατερίνα Κινίτσι. Μας ακούς Κατερίνα, έχεις το λόγο. κυρία Κινίτ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Διευθυντή για την εισήγησή του και επίσης ε, για το έργο που επιτελεί το παρατηρητήριο. Το Ίδρυμα της Ελσαβόνας επιτελεί πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, της πανδημίας, όσον αφορά τα ναρκωτικά. Ίσως αυξήθηκαν αυτοί που απαρτίζουν τα δίκτυα διακίνηση των ναρκωτικών. Επίσης, όπως έγινε και στην κρίση του 2008. Επίσης, ε, τώρα έχουμε διακίνηση πιο επικίνδυνων ναρκωτικών, όπως τότε. Οπότε, για πέστε μας, όσον αφορά το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών, μας είπατε τι γίνεται με τα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης, τι γίνεται με την χρήση στο σπίτι, τι γίνεται από τις σχετικές υπηρεσίες. Από ό,τι φαίνεται, οι τρόποι διακίνησης που υιοθετήθηκαν τώρα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και κόβεται η ομιλήτρια. ancora. Non so ε, Με ακούτε τώρα ξανά συνεχίζει κυρία Κινίτσι. Τι μέτρα χρειάζονται για να μπορέσετε να ε, προσαρμοστείτε όσον αφορά τους νέους τρόπους ε, εμπορίας. Πια αυτά δεν στο δρόμο. Τώρα γίνονται με το ίντερνετ οι κινήσεις των διακινητών. Επίσης κάτι άλλο οι υπηρεσίες σχετικές με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Είπαμε τι γίνεται για αυτή την περίοδο, αλλά μας είπατε και για νέους τρόπους που υπάρχουν όσον αφορά ε, την απαραίτητη θεραπεία. Με βίντεο, με τηλεγιατρική. Επομένως θεωρείτε ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη γι' αυτό τώρα, κάτι τελευταίο για όσα μας είπατε μας είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς πόροι. Είναι σημαντικό για να λειτουργήσει το παρατήριο που μας βοηθάει και εμάς και τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουμε το εμπόριο των ναρκωτικών. Grazie, Εμεί ευχαριστούμε, κυρία Κινίτσι. Ε, και μετά την κυρία Κινίτσι είναι η κυρία Ινετφέλτ για το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Χόρντελ για τα όσα μας παρουσίασε. Και μπράβο του που τα κατάφερε τόσο γρήγορα να συντάξει αυτή την παρουσίαση. Είπαμε ότι υπάρχει μια μετακίνηση, μια αλλαγή από την ποινικοποίηση στην βοήθεια των χρηστών ναρκωτικών. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είπατε ότι ενώ τα κέντρα θεραπείας έχουν πρόβλημα γιατί δεν έλαβαν προστατευτικό υλικό εγκαίρως, αυτό ήταν μια παράληψη. Είπατε όμως ότι έχουμε νέους τρόπους που επινοήθηκαν για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η στροφή από την ποινικοποίηση στην βοήθεια. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμη πολλοί δεν το δέχονται αυτό. Πάντως, επί δεκαετίες, ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών έχει κοστίσει σε χρήμα, σε ζωές και δεν μειώθηκε το εμπόριο. Ακόμα και τώρα με την κρίση δεν μειώθηκε η σχετική δραστηριότητα. Βρέθηκαν άλλοι τρόποι. Επίσης, προβλέπεται ότι Πρόκειται οι έμποροι να βρουν νέες αγορές, νέους τρόπους, περισσότερη βία θα υπάρξει, περισσότερος ανταγωνισμός. Θεωρείτε ότι η παραδοσιακή προσέγγιση θα βοηθήσει. Πεςτε με δύο λόγια παραπάνω. Thank you, Mrs. Now we move Ευχαριστούμε κυρία Ινετφέλντ. Τώρα περνάμε στην ομάδα ID. κυρία Καρδίνο, Ταρντίνο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Διευθυντή. Η σημερινή σας ε, παρουσίαση αφορά την ε, μελέτη που κάνατε σε συνεργασία με την Europol. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ανισχυτικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα καταγράφεται μια σημαντική αύξηση των πώληση ε, των ναρκωτικών στο διαδίκτυο και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες ε, για αυτό το θέμα, μεταξύ των οποίων και το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό οι αστυνομικέ αρχές. Δεύτερον, θα ήθελα να αφερθώ στις συνέπειες της οικονομικής ε, κρίσης. Έχουμε δηλαδή το γεγονός ότι είχαν φοβερές συνέπειες οι μικρές ε, επιχειρήσεις ε, και το θέμα είναι αν μπόρεσαν, αν αναζήτησαν ρευστότητα από ανθρώπους οι οποίοι σε παράνομες δραστηριότητες Επίσης είναι σαφές ότι οι ανήλικοι είχαν περισσότερη διαθεσιμότητα ε, χρήματος. Με αυτό το δεδομένο θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε σε αύξηση φαινομένων όπως οι εκλοπές και οι ληστείες. Επίσης ε, παρατηρήσατε κάποιες ε, συνέπειες όσον αφορά την αύξηση των περιπτώσεων υπερβολικής δόσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους τώρα η κυρία Στρίκ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκόστελ για την έκθεση και την παρουσίαση. Και συμφωνώ με την εκτίμησή του και την ευγνωμοσύνη του για όλο το προσωπικό εκείνο το οποίο εκτέθηκε και χωρί μέτρα προστασία για να βοηθήσει τον άνθρωπο και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Έχουμε ξανά τέτοια υγειονομική κρίση. Επίση ο κ. Χόστελ αναφέρθηκε σε βέλτιστες πρακτικές σε τοπικό επίπεδο όπου υπήρξε επαφή αν ε, υπήρξε επαρκή φροντίδα για τους ανθρώπους και σε κάποια κράτη-μέλη αν υπήρξαν ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ε, δουλειάς τους και πώς θα διασφαλίσετε ότι όντως θα αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα και ότι θα αλλάξουν οι συστάσεις ε, και τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουν οι αρχές. Και τέλος αυτό ίσως σχετίζεται και με την αλλαγή την οποία παρατηρήσατε από την ε, καταστολή, στην φροντίδα και την στήριξη ότι τώρα υπάρχει ε, η ιδέα ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην στήριξη. Ε, και το ερώτημά μου είναι το τι σημαίνει αυτό για τις εθνικές πολιτικές αλλά και για τις πολιτικές της Ένωσης και ίσως και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ίσως θα μπορούσατε να επεκταθείτε σε αυτό γιατί ο πόλεμος ε, των ε, κατά ε, δεν ήταν αποτελεσματικός και κοστίζει πολλά λεφτά. Θεωρείται ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην νόμιμοποίηση αλλά με επένδυση σε πληροφόρηση, φροντίδα και άλλους τρόπους στήριξης. Θα ήθελα την άποψή σας από αυτού και τέλος όσον αφορά την επαφή με τους ανθρώπους. Βεβαίως είναι δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με άτομα τα οποία είναι ήδη περιθωριοποιημένα τι αναμένεται από το προσεχές μέλλον ε, και όταν τελειώσει η καραντίνα. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι φιλοξενούνται σε κοιτώνες ε, και τοπικούς κοιτώνες. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εγκαταληφθούν ξανά και Βεβαίω είχαμε και αυτήν την καινοτομία που αναφέρατε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καταλληλή για όλα τα ευάλωτα άτομα. Πώς θα γεμίσουμε λοιπόν και αυτό το κενό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα για το ECR. Ο κύριος Τσάρλι Βάιμερς. Ε, ε, δεν είναι συνδεδεμένος. με ενημερώνουν ότι δεν είναι συνδεδεμένος. Περνάμε στην Google λοιπόν. Στον πρώτο γύρο πριν ε, ξαναδώσουμε τον λόγο στον διευθυντή. Έχουμε τον κύριο Αρβανίτη από την ΚΟΕ. Είστε συνδεδεμένος, έχετε τον λόγο. Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και που σας βλέπω. Θέλω να πω καταρχήν από την εμπειρία που έχω 30 χρόνια στις θεραπευτικές κοινότητες μην κάνουμε το λάθος ε, για, το, για την ιστορία της καταστολής αλλά και για το θέμα της μικρότερης βλάβης των ουσιών. Οι χρήστες όταν δεν βρουν αυτή την ουσία θα ψάξουν να βρουν μια άλλη ουσία. Ο πόνος προκαλεί χρήση και η χρήση προκαλεί μέγιστο πόνο σε ό,τι αφορά στο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, επιτρέψτε μου να, πω, να ξεκινήσω συγχαίροντα το παρατηρητήριο, το συντάκτη τη έκθεση. Ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο, μια υπέροχη δουλειά, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε όλη την εξαιρετική πορεία που κάνει το παρατηρητήριο για τη δουλειά μα. Θέλοντα να συμβάλλω στη συζήτηση, θέλω να εισφέρω τα εξή. Όπω είναι γνωστό σε όλου μα, στον ΟΗΕ, στο παρατηρητήριο παντού, η αντιμετώπιση των ουσιών που αποτελούν σύνθετο φαινόμενο προϋποθέτει παρεμβάσεις όχι μόνο στο πεδίο της προσφοράς, αλλά και στο πεδίο της ζήτησης. Η ζήτηση επίσης είναι ένα θέμα σύνθετο που εξαρτάται από παραμέτρους όχι μόνο ιατρικές, επιμένω σε αυτό, αλλά και ψυχολογικές και κοινωνικές και πολιτικές σε έναν βαθμό. Ευνόητο είναι ότι οι ίδιες αυτές παράμετροι είναι κρίσιμες για την πολιτική της ανάσχεσης και της θεραπείας του φαινομένου. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς είναι αδύνατο να κάνουμε κατασταλαγμένα στοιχεία για το ψυχολογικό και για το κοινωνικό πεδίο. Η πανδημία του COVID έφερε ήδη σημαντικέ αλλαγέ. Το βλέπω στην πόλη μου, στην Αθήνα, στι κοινωνικέ σχέσει, με την απομόνωση ανθρώπων, καθώ και με τον ψυχισμό του. Αυτέ οι επιδράσει ασφαλώ δεν θα χαθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα αφήσουν, θα λέγα, ένα ίχνο. Θα είναι ίχνο στι πτυχέ των ανθρώπων και στη ζωή του. Η ευρωπαϊκή κοινότητα, τα κράτη-μέλη, οι γειτονιέ θα πρέπει να στηριχθούν σε επιτυχημένε έω τώρα εμπειρίε, όπω είναι αυτέ των θεραπευτικών κοινοτήτων, προκειμένου αξιολογώντα τα νέα δεδομένα να εισφέρουν λύσει και να προωθήσουν πολιτικέ κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων και όχι απομόνωση ή αποκλεισμού. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον ε, πρόεδρο του παρατηρητηρίου, που χαίρομαι που τον βλέπω. Δεν θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με εργαλείο και δικό σας αυτή εδώ την Επιτροπή που συμβάλλει κατά τη γνώμη με τη σκέψη να πούμε πιο δυναμικά σε μια ε, έλεγα ενιαία πολιτική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Arvanitis. Ευχαριστούμε κύριε Αρβανίτη. Ολοκληρώθηκε έτσι ο πρώτος κύκλος ομιλητών. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τον ε, διευθυντή, τον κύριο Χωστέλ, να απαντήσει για 10 λεπτά για να έχουμε μετά και άλλο χρόνο για να κάνουμε ένα δεύτερο κύριο και να επανέλθουμε σε σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και να απαντήσω στις ερωτήσεις των βουλευτών. Πρώτα απ' όλα για αυτό το οποίο ρώτησε η κυρία Αντίπων την οποία ευχαριστώ. Όσον αφορά τις ροές ναρκωτικών ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα, δεν είμαστε σε θέση να μετρήσουμε ε, τον αντίκτυπο. Και βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε σε συνεργασία με τη Europol. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εδώ πέρα και το δίκτυο Retox των σημείων έπαφης που κάνουν ε, φανταστική δουλειά και κάποιοι από αυτούς ε, βεβαίως υποφέρουν και από χρηματοδότηση. Ε, η πανδημία όμως έδειξε ότι κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ωφεληθούν πολύ περισσότερο και στο εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά λοιπόν τις ροές, είναι δύσκολο να το μετρήσουμε. Είχαμε όμως σημαντικές συλλήψεις, ε, κοκαίνης παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Αμβέρσας. Θα έλεγα ότι όσον αφορά την μελλοντική συνεργασία έχουμε εξαιρετικά δεδομένα όσον αφορά την κατάσταση π.χ. στο λιμάνι της Αμβέρσας και στο μέλλον το μέλλον σημαίνει αν έχουμε αρκετά χρήματα για να διατηρήσουμε την ίδια ομάδα ε, θα ωφεληθούμε από την ίδια ποιότητα και ποσότητα ε, πληροφοριών και από άλλα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Ε, θεωρούμε ότι είχαμε μεγάλες συλλήψεις ναρκωτικών την ίδια περίοδο. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι έχει σταματήσει το εμπόριο. Αντιθέτως, μια θετική ε, συνέπεια όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών είναι ότι λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια πιθανώς ε, η διακίνηση η οδική μεταφέρθηκε εν μέρη την θαλάσσια μεταφορά και αυτό πρέπει να το δούμε. Αναφέρατε το γεγονό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και το σκοτεινό διαδίκτυο για την αγορά ναρκωτικών και αυτό το οποίο παρατηρήσαμε από την ανάλυση κάποιων τέτοιων ιστοσελίδων βλέπουμε ότι υπήρξε μια σημαντική μείωση των μεγάλων ποσοτήτων και αύξηση στην πώληση μικροποσοτήτων. Αυτό οφείλεται μάλλον στην πρόκληση της απαγόρευσης κυκλοφορίας που παρέλυσε τις τοπικές παραδόσεις, οπότε αναζητήθηκαν νέες μέθοδοι. Και βεβαίως συνεργαζόμαστε με την Europol η Europol έχει ένα ειδικό κέντρο που ασχολείται με το κυβερνό έγκλημα. Η ανάπτυξη ε, λογισμικού δεν είναι τόσο εύκολη, γι' αυτό συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Europol, αλλά και με το κοινό κέντρο έρευνας της Κομισιόν. Τέλος. Αναφερθήκατε στην βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και μεταξύ των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Συνεχίζεται αυτή και υπάρχουν ενδείξεις ότι σε κάποιες χώρες ίσως αυξήθηκε ειδικά για τον έλεγχο των τοπικών αγορών. Σε αυτή την φάση, εάν δείτε την έκθεση για την αγορά ναρκωτικών που έχουμε συντάξει μαζί με την Europol, έχουμε δημοσιεύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα Δυστυχώς αφορά μόνο όμω ε, τρει ε, χώρε η μελέτη αυτή. Εάν λοιπόν θα υπάρξει μια απόφαση για αλλαγή της εντολής ε, της υπηρεσίας μας, οπωσδήποτε θα θέλαμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό για να κάνουμε έρευνα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο βεβαίως να δούμε ποια είναι η κατάσταση γιατί είναι δύσκολο να μετρήσουμε. Τώρα, έχουμε τα ερωτήματα της κυρίας Κινίτση, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξη της και για την επίσκεψη. Ναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχει γενικός ένας ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτό ε, το οποίο περιγράψαμε με την Europol για την COVID είναι ότι όπως και στην κανονική οικονομία είχαμε μία όθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η οθέτησή του και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από τον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και γενικότερα στην κοινωνία. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούν και τα προγράμματα έλλειψη, ε, πρόληψης και θεραπείας και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. Και έχουμε κάποιες νέες πρωτοβουλίες ε, στο επίπεδό μας για να δούμε ποιες είναι οι νέες εμπειρίες που θα είναι ενδιαφέρουσες ε, για να διδαχθούν τα κράτη μελή Αναφέρατε ε, και εσείς και άλλοι συνάδελφοι τις νέες μορφές ε, θεραπείας, όπως και η κυρία Ινετφέλτ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν και υπάρχουν πολλά. Κυρίως σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Σε κάποιες χώρες, είναι γνωστό εδώ και 10, 15, 20 χρόνια, πως η μεθαδόνη λειτουργεί. Ε, δεν λειτουργεί συστηματικά και με όλους. Ε, πρέπει να γίνει αξιολόγηση και να διασφαλίσουμε ότι αν δεν εφαρμόζονται πολύ αυστηρά κριτήρια, ίσως έχουμε κάποιες άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες ε, και ατυχήματα στο σπίτι και να φτάσει στα χέρια παιδιών. Είναι κάτι που έχει εξολογηθεί λοιπόν σε κάποιες χώρες, όχι παντού. Δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ε, ως κάτι το πανευρωπαϊκό. Αλλά ε, μέρος του προβλήματος ήταν ότι ο κόσμος, ότι, ο κόσμος θεωρεί ότι δεν εμπιστεύεται τους ε, πελάτες. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε δει, έχουμε και διαδικτυακά σεμινάρια, έχουμε και ένα στις 12 η ώρα, μία η ώρα ώρα Βρυξελών, για το θέμα της πρόληψης και του COVID. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι για την ιατρική ομάδα, για τα κέντρα θεραπείας, Κάποιοι ανέφεραν ότι υπήρχε μια συμφωνία κυρίων με τους πελάτες και ότι όταν σταθεροποιούνται ε, με την θεραπεία τους τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον ε, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις καθώς δεν ήταν δυνατόν να μιλήσουν και να συναντήσουν τους ασθενείς κάποιες από τις ε, συνεντεύξεις ε, και τα σχετικά έγιναν με τηλέφωνο ή και με τηλεδιάσκεψη σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα υποκαταστήσει την θεραπεία, αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο πριν από πέντε μήνες θα απέριπταν οι περισσότεροι γιατροί. Ε, τώρα είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίω δεν είναι το ίδιο και δεν μπορεί να γίνει η ίδια δουλειά αλλά διατηρείται έτσι μια σχέση με τους ασθενείς εκείνους που χρειάζονται κάτι παραπάνω. Και βεβαίως για το πώς θα δοθεί περισσότερη στήριξη στο παρατηρητήριο. Πρώτα απ' όλα ε, χρειάζεται ένας επαρκής προϋπολογισμός για το 2021 ως αφετηρία για το επόμενο ΠΔΠ και το δεύτερο και ήδη έχουμε περάσει την εποχή μετά τον COVID για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας η Κομισιόν. Έχει, ανακοινώσει, έχει κάνει μια ανακοίνωση για την εξωτερική αξιολόγηση του κέντρου. Υπάρχουν κάποιες ιδέες και κάποιες ανάγκες και ευκαιρίε ε, που έχουμε ταυτοποιήσει για να διευρυνθεί η εντολή μας, για να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι φέτος έχουμε τα 25 χρόνια της παρακολούθησης, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια και πολύ περισσότερα τους τελευταίους πέντε μήνες. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την υπηρεσία αυτή στις νέες εποχές. Για την κυρία Ενετφέλ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην πράξη Για μένα ένα από τα διδάγματα της κατάστασης είναι ότι οι γιατροί, οι τοπικές ομάδες, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, είναι σε επαφή με, και αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Και βεβαίω αυτό έχει γίνει με ρεαλισμό, όχι με δόγμα. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή. Δεν εμπιστευόμαστε τους χρήστες γιατί είναι αφελείς κτλ. Όχι, αν είναι οι πελάτες μου, έχουν δυσκολίες να επιζήσουν και πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί δεν μπορούμε να τους ε, υποδεχόμαστε κάθε μέρα ως συνήθως. Και είναι δύσκολη κατάσταση γιατί μπορεί να έχουν εκτεθεί στον COVID και αυτή και το προσωπικό. Βεβαίω αυτό σχετίζεται και με την εθνική νομοθεσία. Σε κάποια περιπτώσει, παραδείγματο χάρη, δεν προβλέπει η νομοθεσία να παίρνουν μεθαδόνη στο σπίτι και αυτό θα απαιτήσει κάποιες ε, νομοθετικές αλλαγές. Αλλά οι γιατροί μας είπαν ε, και αυτό έγινε και στο σεμινάριο ότι αυτά είναι κάποια από τα ωφέλη χρηστών και επαγγελματιών ότι πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία πριν από πέντε μήνες θεωρούσαμε ότι δεν ήταν ε, δυνατά να γίνουν, αλλά πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση. Και επειδή υπάρχει και το θέμα του χρόνου, θα απαντήσω μαζί στις ερωτήσεις ε, των κυρίων Ταλντίνο Στρίκ και του κυρίου Αρβανίτη. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ερώτηση ήταν η εξής. Αυτό το οποίο ακούμε κάθε μέρα, πώς μπορούμε να στηρίξουμε ε, την λήψη αποφάσεων καλύτερα. Πώς θα φροντίσουμε δηλαδή να λύσουμε διδάγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ξεκινήσει πολλές νέες πρωτοβουλίες ε, σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό κτλ. Και με αυτούς που ασχολούνται με τη θεραπεία. Είμαστε σε τηλεδιάσκεψη με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον έλεγχο των ασθενειών και θα παρουσιάσουμε κάποιες αναλύσεις και εκθέσεις για τον αντίκτυπο του COVID και τη διαχείρισή του. Γιατί εδώ βεβαίω βλέπουμε το πώς έγινε η διαχείριση της πανδημίας και θα ήθελα εδώ πέρα να στηρίξω τον ρόλο της αδελφής μας υπηρεσίας του ECDC του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών και νομίζω καλό είναι να σταματήσουμε να χτυπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και εμείς και το ECDC και η Europol είχαμε αποτελέσματα 24 ώρες το 24ωρο και νομίζω καλό είναι να δοθεί η δημοσιότητα που αξίζει σε αυτό. Και τέλος, για τις ευκαιρίες μελλοντική ε, παρακολούθησης. Νομίζω πως γίνεται ενδιαφέρουσα δουλειά αυτή τη στιγμή. Είχαμε την αξιολόγηση της τελευταίας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Κομισιόν προετοιμάζει τα επόμενα βήματα και βεβαίως όλα αυτά τα διδάγματα θα μας καθοδηγήσουν και στο μέλλον και βεβαίως ε, και εμείς ε, παρέχουμε όλη την στήριξη των κομισιών και στις επιτροπές του Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή σας ε, και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και βεβαίως στην ομάδα για το πρόγραμμα Horizon. Βεβαίως, Ένα λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η έκθεση από κοινού με την Europol είναι ότι εμείς και η Europol θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εικονική διάσκεψη που θα λάβει χώρα στις 26 Ιουνίου και θα παρουσιάσουμε αυτήν την έκθεση με, τα, με τις τελικές παρατηρήσεις μας βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις αυτές που μας δώσατε και για τα θέματα αυτά τα οποία ανέφεραν οι ομιλητέ στον πρώτο γύρο. Έχουμε το δεύτερο γύρο και έχουμε κάποια μέλη τα οποία θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα πρότεινα λοιπόν τώρα να του δώσουμε το λόγο για να μας κάνουν τι ερωτήσεις τους. Ο κύριος Πίκερς, πρόσωπο του ΕΛΚ. Αν μας ακούτε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Πίτερς ε, έφυγε. Ο κύριος Πίτερς λοιπόν δεν είναι παρόν. Η κυρία Σίπελ. Για αυτή ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Κουζδέλ. Και να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι πολλά σημαντικά ερωτήματα ήδη έχουν απαντηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε δύο μόνο σημεία και θα συνεχίσω στα γερμανικά, αν με επιτρέπετε. Σκεφτόμενοι αυτούς που καταναλώνουν ναρκωτικά, θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι είναι εξαρτημένοι και παίρνουν ανατακτικά ναρκωτικά και κατά τα άλλα έχουν μία λίγο πολύ ρυθμισμένη ζωή και οι άλλοι που ζουν στον δρόμο. Έχετε λοιπόν αποτελέσματα ακόμα και αν συνεχίζετε η κατανάλωση των ναρκωτικών χωρίς ε, μεγάλες αλλαγέ, κατά πόσον αυτέ οι δύο ανθρές κατηγορίες ε, έχουν κάποιε διαφορέ να επιδείξουν κατά πόσον υπάρχει μια μεταβατική φάση, ψυχολογικά προβλήματα, ενδεχομένω αν υπάρχουν τάσεις βίας στις οικογένειές τους και το καθεξής. Και μια ερώτηση ακόμα για την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα μεθαδόνης, όπου υφίστανται αυτά. Εξ όσων κατάλαβα, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Γιατί ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον έχετε συμπεράσματα σε περιπτώσεις όπου δεν συνεχίστηκε η παροχή μεθαδόνης για θεραπευτικούς σκοπούς, κατά πόσον αυτό ενδεχομένως προκάλεσε αλλαγή χρήση ναρκωτικών, αλλαγή είδου χρήση, δηλαδή. Και τώρα δηλαδή κατέληξαν οι άνθρωποι αυτοί να χρησιμοποιούν και πάλι άλλε άλλες Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και ο Ευχαριστούμε την κυρία Σίπελ. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Μια και ο κύριο Πίτερ ε, αποχώρησε, η κυρία Σίπελ πήρε το λόγο. Δεν έχουμε άλλον βουλευτή στην αίθουσα ή μέσω σύνδεση που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Άρα να δώσουμε το λόγο πάλι στον κύριο Κουζτέλ για να κάνει κρατικά σχόλια για το θέμα αυτό. Έχετε και πάλι το λόγο λοιπόν. Παρακαλώ πιέστε το πλήκτρο speak. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Σίπελ για την ερώτηση αυτή και για τα σχόλια που κάνετε Για την πρώτη ερώτηση τώρα. Ναι, φυσικά. Έχουμε διάφορες κατηγορίες και προφίλ χρηστών. Και έχετε δίκιο που αναφέρετε ότι κάποιοι εξ αυτών ή μάλλον πολλοί εξ αυτών έχουν κοινωνική ένταξη σε έναν βαθμό δεν μιλάμε μόνο για την ε, καρικατούρα του Τζάνκι που είχαμε υπόψη μας στα τέλη της δεκαετίας του 80. Φυσικά υπάρχουν και πιο ευάλωτοι άνθρωποι. Αλλά έχουμε άτομα τα οποία έχουν λίγο πολύ μια σταθερή θεραπεία και θυμάμαι ότι κάποιοι από τους συναδέλφους μας έκαναν μια παρατήρηση ότι ενδεχομένως να μην υπάρχουν δυνατότητες τηλεθεραπείας, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλισέ δεν είναι το ίδιο. Η πραγματικότητα μάλλον δεν ανταποκρίνεται στο κλισέ που είχαμε πριν από 30 χρόνια. Έχουμε μετά και τα άτομα τα αυτά που έχουν πολλούς παράγοντες ευαλωτότητας, συγκεντρωμένους. Ένα θέμα είναι ότι σήμερα οι γυναίκε οι οποίε χρησιμοποιούν ναρκωτικά είναι ακόμα στιγματισμένε. Αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση. Και συχνά δεν υπάρχει σωστή παροχή θεραπεία η οποία να συνάντηκε με τι ε, ανάγκε του. Για όλα λοιπόν αυτά τα άτομα έχουμε διαφορετικούς, ε, διαφορετικές συνθήκες. Και σήμερα είναι δύσκολο να μετρήσουμε τον αντίκτυπο. Αυτό που ξέρουμε και αυτό επιβεβαιώθηκε άλλωστε και στο πρώτο webinar για τον αντίκτυπο του COVID στις θεραπείες είναι ότι τα προγράμματα και τα κέντρα θεραπείας πραγματικά χρειάζεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Αλλά το θέμα δεν ήταν μόνο να χορηγούνται σύριγγες ή να δίνεται πληροφορίε για τις θεραπείες. Χρειάζονταν και βασικό εξοπλισμό οι άνθρωποι αυτοί και έπρεπε να τους χορηγηθεί. Και άρα, από αυτή την άποψη, το Μάρτιο και όταν λάβαμε ε, σχόλια και ερωτήσεις από τους συναδέλφους, αισθάνθηκα και πάλι όπως στην αρχή της δεκαετίας του 90. Στην Γαλλία υπήρχε μια οργάνωση που ονομαζόταν Λίμι Τελακάς. Η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη από την επιδημία του HIV και του AIDS που είχε προκληθεί πανικός παντού. Ιδιαίτερα για αυτούς που είχαν μεγαλύτερη έκθεση. Αλλά όπως σας είπα, Παρ' αυτά, σε κάποιες χώρες ήταν δυνατόν να συζητηθούν και να βρεθούν πόροι. Σε τελική λοιπόν ανάλυση, σκοπός μας ήταν να περιορίσουμε αυτό που αναφέρατε δικαίως, τις ε, μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες των προγραμμάτων. Τώρα, για τη δεύτερη ερώτηση. Νομίζω ότι βάσει αυτών που λάβαμε ως τώρα, ως στοιχεία, δεν έχουμε λάβει ουσιαστικά πληροφορίες ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με άτομα τα οποία ενδεχομένω να βγαίνουν από τα προγράμματα χρήση μεθαδόνης. Ενδεχομένω να υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες χώρες. Γιατί, για παράδειγμα, κλείσαν τα κέντρα παροχής μεθαδόνης ή ενδεχομένως να λειτουργούσαν ε, πιο περιορισμένες ώρες. Από την Ιταλία μας ε, είπαν κάποιοι χρήστες ότι ένα από τα πρώτα μαθήματα τα οποία έμαθαν ήταν ότι σε μελλοντική επιδημία θα πρέπει να διευρύνουν το ωράριο εργασίας, όχι να το βραχύνουν, γιατί σε περίπτωση επιδημίας υπάρχει λιγότερη συγκέντρωση χρηστών αν υπάρχουν πιο ευρεία ωράρια. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία για άτομα τα οποία έχουν εγκαταλείψει τα πρόγραμματα α, παροχής υποκαταστατών ουσιών. Αλλά μία από τις προκλήσεις για τις οποίες δεν έχουμε ακόμα σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά ήδη νωρίς, το Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, λάβαμε αιτήματα για πληροφορίες από πρόγραμματα θεραπείας σε τρία-τέσσερα τουλάχιστον κράτη-μέλη που μας είπαν ότι ε, κοιτάξτε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε άτομα τα οποία χρησιμοποιούν οπιοειδή και δεν ε, μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στα, στις ουσίες αυτές. Ή έχουν ε, ουσίες πολύ χαμηλής ποιότητος ή υποκαθιστούν τις ουσίες αυτές με ακόμα πιο επικίνδυνες ουσίες. Κάποιοι εξ αυτών ε, δεν μπόρεσαν να αντέξουν ε, τη στέρηση. Και το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια κρατημέλη τουλάχιστον οι συνθήκες για την αξιολόγηση του ασθενή πρωτού του επιτραπεί να μπει σε πρόγραμμα μεθαδόνης και κατά πόσον είναι κατάλληλος ε, για τη χρήση υποκατάστατου και τη δοσολογία θα χρειαζόταν. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπόρεσαν να γίνουν πλέον. Και οι δυσκολίε λοιπόν ήταν αυτές. Ε. Κατά πόσον υπήρχαν ε, επίσης ε, εμπειρίες από άλλα Βρήκαμε λοιπόν τέτοιες εμπειρίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα παράδειγμα καλής πρόοδου. Προφανώς πρέπει να ορίζονται και οι όροι, γιατί προφανώ πρόκειται για κλινική χρήση. Δεν είναι εμπορική η χρήση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι ο ασθενή θα ωφεληθεί από την θεραπεία και δεν θα υπάρξουν παράπλευρε ε, συνέπειες. Κίνδυνο, για παράδειγμα, υπερβολικής χρήση. Για το σχόλιο του κ. Αρβανίτη, για να απαντήσω και στην κυρία Ιντφέλντ. Ένα ποίημα του Καβάφη, της Ιθάκης του Καβάφη. Το μυθικό, περίφημο ποίημα. Οι λεστριγόνες, οι κύκλοπες, τα τέρατα λοιπόν αυτά. Όταν τους απαντάς, δεν μπορείς να τους απαντήσεις, εκτός και να τους φέρεις στην ψυχή σου. Νομίζω ότι οι επαγγελματίε του κλάδου, η κοινωνική λειτουργία κτλ. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τι αποφάσει, μα είπαν ότι αυτό που ουσιαστικά αποτρέπει την ε, λήψη αποφάσεων είναι οι εσωτερικές ε, προκαταλήψεις που έχουμε ο καθένας μας. Και να πω ότι πέρα από τις ελλείψεις αυτές και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ελπίζω να σας έδειξα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε θέματα σε ό,τι αφορά τη μείωση παροχής ζήτησης, σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες ε, των ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μοναδικό μοντέλο στον κόσμο αυτό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σώζει οι ζωέ. Λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα παλιά μέτρα. Τελικά, να μην είναι αυτοί που αποφασίζουν για το θέμα αυτό και οι χρήστε οι οποίε θα πληχθούν και την δεύτερη φορά. Χρειάζεται λοιπόν ε, προετοιμασία, παρέμβαση για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας. Και τους τελευταίους μήνες υπήρξε αύξηση στην παροχή ναρκωτικών. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα συνεχιστεί ο στάση για κάποιες από τις ουσίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα ναρκωτικά ε, δεν πρόκειται να πάψουν να υπάρχουν. Θα είναι τμήμα μιας μελλοντικής ε, επιδημίας. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε. Όχι να μειώσουμε του προπολογισμού και να πούμε σε τρία-τέσσερα χρόνια ότι α, μήπω θα πρέπει κάτι να επενδύσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να προετοιμαστούμε εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χοστέλ. Ευχαριστούμε για όσα μας ε, εξηγήσατε. Σας προσέξαμε, σας παρακολουθήσαμε σε όλα τα ζητήματα που καλύψατε από όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε και εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο της υπηρεσίας σας. Επίσης, ε, βεβαίως και θα λάβουμε υπόψη το θέμα το οικονομικό, το δημοσιονομικό που είπατε για τη χρηματοδότηση της ε, υπηρεσίας σας. Ε, ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Επίσης, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημέρα σε διάταξη. Τα καταφέραμε, ολοκληρώσαμε πριν το προβλεπόμενο χρονικό όριο και έτσι εξαντλήθηκε η μερική Αλλά πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, την σημερινή, ε, σας λέω θα τα ξαναπούμε το απόγευμα. Ε, θα ξεκινήσουμε στις 4 ε, και 4. Πρώτα πρώτα έχουμε το σχέδιο έκθεσης της Νομικής Επιτροπής για το ζήτημα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Σας θυμίζω ότι έχουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που είναι η 11η Ιουνίου. Κάτι σας είπα και η κυρία Κιάνκο. Στις 4 η ώρα. 11 4 το απόγευμα. Επίσης κάτι άλλο που θα σας πω είναι το εξής, ότι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα σας στείλουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Schengen σε σχέση με την πανδημία. Αυτά. Το απόγευμα, το απόγευμα στις 4 και 50 θα τα ξαναπούμε, αλλά θα σας στείλουμε ένα email. Και